Δεν ξέρω αν ε, θα ε, είμαστε ε, τόσοι διότι δεν κατορθώσαμε να ακολουθήσουμε το χρόνο στην κοινή συνάντηση που είχαμε με την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Θα πρότεινα λοιπόν να συνεχίσουμε παρόλο που είμαστε λίγοι μέσα στην αίθουσα. Έχουμε λοιπόν προσκαλέσει τον υποψήφιο διευθυντή του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, ETF, ε τον Σεζάριο Νεστίνη και ε, θα ε, ξεκινήσουμε λοιπόν δίνοντας τον λόγο στον κύριο Νεστίνη για την πρώτη του ομιλία και στη συνέχεια τα μέλη θα έχουν την δυνατότητα να θέσουν ερωτήματα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 αξιότιμα μέλη του Κοινοβουλίου. Κυρίες και κύριοι, αποτελεί μεγάλη ευχαρίστηση που βρίσκομαι ανάμεσά σας ε, και ε, μπορώ να σας συστηθώ και να μοιραστώ μαζί σας το όρομα που έχω ε, για τον ρόλο που θέλω να λάβω ως Διευθυντής του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. Πρώτη μου λοιπόν προτεραιότητα θα είναι να δώσω ε, ορατά αποτελέσματα ε, στην εντολή του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματική Εκπαίδευσης, το οποίο είναι να προωθήσει την ε, ανάπτυξη του ανθρωπίνου κεφαλαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως, για να το προωθήσουμε αυτό, το ETF θα πρέπει να κάνει σειρά πραγμάτων, όπως για παράδειγμα να δώσει ειδικευμένη γνώση, τεχνοδοσία και κοινοτόμες ιδέες και δεύτερον θα πρέπει να συνεχίσει να συνεργάζεται και να ενισχύει τις σχέσεις του με τους εταίρους και τέλος θα πρέπει ε, να ε, χρησιμοποιεί ε, ορθά και αποτελεσματικά τους πόρους του. Ε, να ε, αναπτύξω κάποια πράγματα για αυτό και στο τέλος θα πω και ε, κάποια, θέμα, κάποια πράγματα για τον εαυτό μου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ταυτοποιήσει την ανάπτυξη των δεξιοτήτων ως μία από τις πολιτικές της προτεραιότητες που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της προώθησης της κοινωνικής Ευρώπης και σε αυτό το πλαίσιο το ETF καλείται να συνεισφέρει σε αυτή την ατζέντα μοιράζοντα τεχνογνωσία με τους εταίρους και να διασφαλίσει κοινό κέρδος μέσω της συνεργασίας. Η προώθηση η ανάπτυξη του ανθρωπίνου κεφαλαίου συνεισφέρει στην οικονομική ανάπτυξη, την παραγωγικότητα και την απασχολησιμότητα και επιπρόσθετα η ανάπτυξη ανθρώπινου κεφαλαίου σημαίνει ε, ε κοινωνική συνοχή και μεγαλύτερη ενασχόληση με τα κοινά. Συνεισφέρει στην ανάπτυξη και την εφαρμογή το, της πολιτικής εξωτερικών σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρέχοντας ειδικευμένη γνώση στους τομείς της. Ε, στο πλαίσιο της εξωτερικής δράσης η Ευρωπαϊκή Ένωση όπως γνωρίζετε έχει επενδύσει ιδιαίτερως σε στενότερες σχέσεις με τους εταίρους και άλλες χώρες εταίρους που έχουν ε, ταυτοποιηθεί ως ε, συνεργάτες του ETF. Η ανάπτυξη ανθρωπίνου κεφαλαίου λοιπόν είναι αναπόσπαστο κομμάτι της Ευρωπαϊκή Ένωση για να συνεισφέρει στην οικονομική και κοινωνική μεταμόρφωση των χωρών εταίρων και αυτό είναι προ συμφέρον της Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και των χωρών εταίρων για να προωθηθεί σταθερή βιώσιμη ανάπτυξη, ενίσχυση των ε, σχέσεων και κάνοντας αυτό, ε, οι αρχήβα στις οποίες οι δημοκρατικές διαδικασίες εκπορεύονται από τα έθνη ε, είναι υψή της σημασίας. Το αποτέλεσμα λοιπόν είναι σημαντικό για την βιωσιμότητα και την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων μακροπρόθεσμα. Οι παγκόσμιες τάσεις, όπως γνωρίζει αυτή η Επιτροπή, ε, μεταμορφώνουν τις ανάγκες ικανότητες και δεξιότητες. Υπάρχει επίγνωση των κινδύνων ότι ορισμένες χώρες, όπως και ορισμένοι τομείς του πληθυσμού, είναι πιο ευάλωτοι σε τέτοιε αλλαγέ σε περίπτωση που δεν μπορέσουν να προσαρμοστούν. Μέσω του ETF λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να υποστηρίξει χώρε εταίρου ε, για να αντιμετωπίσουν αυτέ τι προκλήσει, να μάθουν ε, ο ένας, η μία χώρα από την άλλη και να ταυτοποιήσουν τι δυνάμει και αδυναμίε του οι ε, προκλήσεις ε, όσον αφορά την προσαρμογή στις ε, βιομηχανικές αλλαγές, η επανεκπαίδευση είναι βασικοί τομείς πάνω στους οποίους εργάζεται το ETF και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αρκετά εργαλεία τα οποία έχουμε αναπτύξει και στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως είναι η κινητικότητα, το πλαίσιο δεξιοτήτων τα οποία μπορούν να μοιραστούν και οι χώρες που συνεργάζονται με το ETF. Επιπρόσθετα, οι χώρες εταίροι έχουν και παρόμοιε προκλήσει αλλά και διαφορετικές ανάγκες και βρίσκονται σε διαφορετικά ε, στάδια στα δικά τους εθνικά πλαίσια ε, προώθησης δεξιοτήτων, διαβίου μάθησης και ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου και γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να αναπτύξουμε εργαλεία για να ανταποκριθούμε σε αυτές τις ανάγκες και το ETF ε, μπορεί να συνεισφέρει σημαντικά σε όλο αυτό και επιπρόσθετα μπορούμε να έχουμε τομεακή προσέγγιση που μπορεί να εφαρμοστεί σε όλες τις χώρες εταίρους. Το ETF ε, ε, θα συνεχίσει να προωθεί το νέο τρόπο σκέψης, ε, να αναζητεί εταιρικέ σχέσεις και να προβλέπει καλύτερα τις ανάγκες του μέλλοντος. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να συνεισφέρουμε στους ευρωπαϊκούς μας στόχους για τη διασφάλιση της σταθερότητας και της ευμάρειας σε αυτά τα μέρη του πλανήτη. Τώρα θα ήθελα να σας πω κάποια πράγματα για τους κυρίους εταίρους που έχουμε. Το ETF ε, συνεχίζει να υποστηρίζει το έργο του ε, σε στενή συνεργασία με τους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, συνεργάζεται με τους θεσμούς αλλά και πέρα από τους θεσμούς με ερευνητικά όργανα και άλλους παγκόσμιους παράγοντες παρέχει εξειδικευμένη γνώση στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε σημαντικά ζητήματα ζητήματα όπως είναι οι δεξιότητες, η εκπαίδευση και η κατάρτιση. Ε, εργαζόμενοι με τα κράτη, συνεργαζόμαστε με τα κράτη-μέλη επίσης και με αυτό τον τρόπο μπορεί να δημιουργήσει συνεργίες με τα κράτη-μέλη το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λοιπόν αποτελεί έναν σημαντικό συνομιλητή ε, του ETF και εγώ ως ε, διευθυντής θα συνεχίσω να το πρώτο αυτό. Η λογοδοσία προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διασφαλίζει ότι το ETF μπορεί να, να παίξει το ρόλο του με κυριότητα, διαφάνεια και υπευθυνότητα και χαιρετίζω τις καλές σχέσεις τις οποίες ανέπτυξε η προκάτοχο μου με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και δεσμεύομαι να συνεχίσω να το κάνω αυτό. κάνοντας ε, το έργο του, το ETF επίσης πρέπει να λειτουργήσει και ως ε, γέφυρα μεταξύ των ε, παραγόντων πέρα από τους θεσμούς και θα συνεργαστούμε βέβαια και με την αδελφή υπηρεσία, την SEDEFOP, όπου απαιτούνται συνεργίες και κοινή προσέγγιση που θα συνεχιστεί με όμοιο τρόπο και με άλλους τομείς. Ένα βασικό συστατικό ε, για το ETF θα είναι να διασφαλίσει ότι η τομή ε, υπευθυνότητα θα είναι να ξεκινήσει διάλογο με τρίτε χώρε, καθώ προσπαθούμε να ενώσουμε του διάφορου ευρωπαϊκού παράγοντε, ούτω ώστε όταν εργαζόμαστε πάνω στου τομεί προώθηση τη ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου σε τρίτε χώρε, ε, θα, θα μπορούμε να ενώνουμε όλου του συνομιλητέ που δουλεύουν πάνω σε αυτή τη χώρα. Μερικέ χώρε υπό την εντολή του ETF αντιμετωπίζουν χτίζουν εσωτερικές εντάσεις, εμφυλίους πολέμους, πολιτικές εντάσεις και προφανώς ε, το ETF πρέπει να θέσει προτεραιότητες στη δράση τους ε, και με το Διοικητικό ε, Συμβούλιο, υπό την καθοδήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι προτεραιότητες αυτές συζητούνται στο πλαίσιο του ετησίου προγράμματος. Όμως η τεχνογνωσία του ETF μπορεί να βοηθήσει ιδιαίτερως ακόμα και χώρες που βιώνουν μεταρρυθμίσεις και σχετικά με ζητήματα τα οποία ε, αφορούν και προκύπτουν όταν ε, αρχίζουν οι χώρες αυτές ε, να αποκαθίστανται και εκεί λοιπόν το ETF παίζει σημαντικό ρόλο σε αυτήν την μεταρρύθμιση αλλά και η χειραφέτηση των γυναικών παίζει ένα σημαντικό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία όπου μπορεί να συνεισφέρει το ETF. Το τελευταίο σημείο το οποίο θα ήθελα να αναφέρω είναι η ε, ορθή και αποτελεσματική διαχείριση των πόρων. Όπως όλοι οι δημόσιοι οργανισμοί που εργάζονται για την Ευρωπαϊκή Ένωση, το ETF θα πρέπει να χρησιμοποιεί τους πόρους του αποτελεσματικά και ως ε, ε, ε, υπηρεσία έχουμε στόχο να αναπτύξουμε το ανθρώπινο κεφάλαιο το οποίο αποτελεί και το βασικό του πόρο. Η τεχνογνωσία που έχει είναι το βασικό της προτέρημα. Σε περίπτωση που γίνω διευθυντής τότε ε, έχω σκοπό να συνεχίσω να εφαρμόζω ε, τους, ε, τις υπάρχουσες μεσοπρόθεσμες προοπτικές εσωτερικές και εξωτερικές αξιολογήσεις έχουν δείξει ότι ε, η υπηρεσία διαχειρίζεται καλά τους πόρους της ε, και οι αξιολογήσεις έχουν δείξει ταυτόχρονα ότι υπάρχουν τομείς ε, όπου απαιτείται περαιτέρω προσοχή και σε αυτούς τους τομείς θα επικεντρωθώ ιδιαιτέρως. Ε, η ε, παροχή ηγεσία και κατεύθυνση στο προσωπικό τη υπηρεσία θα αποτελέσει τον βασικό μου ε, στόχο, διότι μονάχα στην περίπτωση που εργαστούμε ω ομάδα θα μπορέσουμε να επιτύχουμε του στόχου και την εντολή μα. Ω διευθυντή λοιπόν θα λειτουργώ για το γενικό συμφέρον τη Ευελινωσή ύστερα από 22 χρόνια ε, υπηρετώντας τους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεσμεύομαι να προωθήσω τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, είχα ε, την τιμή να εκπροσωπήσω τους τομείς, την Ευρωπαϊκή Ένωση στους τομείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης και εκεί αφιέρωσα τα πρώτα χρόνια της καριέρας μου και είναι τομείς στο πλαίσιο των οποίων εργάστηκα σε, διάφορους, ε, σε διάφορες περιοχές του πλανήτη. Υπηρέτησα την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, με τις ε, αποστολές της στη Νέα Υόρκη αλλά και στην Ινδία και έχω αρχίσει να εκτιμώ το τι είναι οι ευρωπαϊκές αξίες, κάτι το οποίο προωθεί και το ETF και το πόσο σημαντική είναι η δράση που κάνουμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση σε τρίτες χώρες και με βάση αυτές τις αξίες υπόσχομαι να κάνω ό,τι μπορώ για να ε, διασφαλίσω ε, την καλή λειτουργία της υπηρεσίας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Είναι λίγα τα μέλη τα οποία είναι παρόντα. Αλλά ίσως υπάρχουν ερωτήσεις για Ευχαριστώ. Είναι λίγα τα μέλη που είναι παρόντα, αλλά θα συνεχίσουμε με ερωτήσεις για εσάς. Συντονίστρια. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Ονεστίνη για την παρουσίασή σας. Πιστεύω πως το βιογραφικό σας με τόση εμπειρία στις εξωτερικές σχέσεις είναι χρήσιμο για τη θέση που αναλαμβάνετε. Η προκατοχό σας είχε συνεργαστεί πολύ στενά με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ήταν μια πολύ γόνιμη συνεργασία και τις δύο πλευρές, τόσο το ETF όσο και μας στην Επιτροπή μας άρεσε και μπορέσαμε και αποφεληθήκαμε πολύ από αυτήν και ελπίζω η συνεργασία αυτή να συνεχιστεί και μέσα στο Διευθυντή. Τρεις ερωτήσεις έχω προς εσάς, τέσσερις μάλλον. Τα κίνητρά σας να γίνετε Διευθυντής του ETF. Μέχρι στιγμής είχατε πολύ ενδιαφέρουσες θέσεις τι είναι αυτό που σας παρακινεί να γίνετε διευθυντής του ETF. Δεύτερη ερώτηση. Θέλετε νέες εταιρικέ σχέσεις για μελλοντικές ανάγκες. Τι εννοείτε συγκεκριμένα. Τρίτη ερώτηση. Κατά την άποψή σας, ποιες είναι οι σημαντικότερες προκλήσεις για την πολιτική, όχι για την υπηρεσία, για την πολιτική τα επόμενα χρόνια και αυτό που μου λείπει λίγο και οι συνάδελφοι γνωρίζουν πως ασχολούμαι με αυτό ιδιαίτερα είναι η ψηφιοποίηση. Αυτές είναι οι ερωτήσεις μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσίασή σας. Παρακαλώ κύριε Νεστίνη. Σας ευχαριστώ για τις ερωτήσεις. Με ρωτήσατε για το κίνητρό μου. Πιστεύω ακραδάντως και αυτό κινητοποίησε την ε, δράση μου αυτή, ότι η εκπαίδευση και η κατάρτιση βρίσκεται στο επίκεντρο των μετασχηματισμών της κοινωνίας. Είναι μεγάλη πρόκληση να κομίσουμε εμπειρογνωμοσύνη σε τρίτες χώρες που είναι τόσο σημαντικοί εταίροι της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουμε το κίνητρο να συνδυάσουμε τις δεξιότητες που έχουν να κάνουν και με το ε, σκέλος των εξωτερικών σχέσεων. Έχω εργαστεί σε θέματα εξωτερικών σχέσεων και σχέσεων με τρίτες χώρες και έχω εμπειρογνωμοσύνη να κομίσω. Και θέλω αυτή, αυτές τις γνώσεις να τις συνδυάσω ε, με τις γνώσεις για την ε, επαγγελματική εκπαίδευση, για την κατάρτιση μεταξύ άλλων. Η γειτονία μας είναι η πιο σημαντική από τις πιο σημαντικές πολιτικά για την ε, ευρύτερη ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό το είδαμε και με τα πρόσφατα γεγονότα. Είδαμε πόσο σημαντική είναι η πρόθεση της σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή. Αυτό είναι κάτι που ενδιαφέρει άμεσα και τους Ευρωπαίους καθεαυτούς. Είδαμε το κόστος και το κίνδυνο της αστάθειας, πόσο μεγάλα είναι. Γνωρίζουμε ότι είναι κοινό συμφέρον να προωθήσουμε τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή, στη γειτονιά μας. Θέλω όλες τις εμπειρίες που έχω συλλέξει όλα αυτά τα χρόνια, από όλα τα μετερίζια στα οποία έχω υπηρετήσει, να τα συνδυάσω σε αυτό το τομέα εξέχουσας πολιτικής σημασίας που είναι η ανάπτυξη του ανθρωπίνου κεφαλαίου. Ω προ τι εταιρικέ σχέσει, θεωρώ ότι το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα επαγγελματική εκπαίδευση μπορεί να διαδραματίσει το ρόλο που του αναλογεί μόνο αν βρίσκεται στο επίκεντρο ενό ισχυρού δικτύου παραγόντων και δρόντων φορέων. Παρέχει αναλύσει, εμπειρογνωμοσύνη, γνώσεις, ειδικότητα, αλλά οι εθνικέ αρχέ θα αξιοποιήσουν τα κοινοτικά προγράμματα και θα δημιουργήσουν παραδοτέα. Και υπ' αυτή την έννοια θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντική η εταιρική σχέση μέσα από τα διάφορα τμήματα, με τα διάφορα τμήματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αλλά και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μόνο έτσι μπορούμε να φέρουμε αποτελέσματα. Άρα βασική μας ιδέα δεν είναι να αναπτύξουμε νέες εταιρικές σχέσεις, αλλά να ενισχύσουμε τις θεσμικές διασυνδέσεις. Τη σύνδεση του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης με τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό να τυποποιηθεί, να γίνει καθεστώς ως προς τον τρόπο με τον οποίο φέρνει αποτελέσματα το Ευρωπαϊκό αυτό Ίδρυμα. Είναι δύσκολο βέβαια να σας δώσω απάντηση με δύο λόγια ε, σε σχέση με το επόμενο ερώτημά σας. Ωστόσο, μιλώντας για τις αρμοδιότητες του Ιδρύματος αλλά και τη γεωγραφική του αρμοδιότητα, θεωρώ ότι συλλογικά η πρόκληση που μας απασχολεί είναι το πώς θα ανταποκριθούμε και ποια αντίδραση θα επιφυλάξουμε στην παγκοσμιοποίηση, πώς θα δράσουμε ε, έναντι του μετασχηματισμού του χώρου της εργασίας ε, και των θέσεων απασχόλησης, ο οποίος προκαλείται από την παγκοσμιοποίηση. Βλέπουμε την απάντηση που επιθυμεί να δώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην πολιτική της ατζέντα. Όλα αυτά είναι προτεραιότητες εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι και στοιχεία κλειδιά που θα πρέπει να διέπουν τις σχέσεις μας με τις γειτονικές χώρες. Επομένως, πώς θα αντιδράσουμε στην παγκοσμιοποίηση, πώς θα έχουμε θέσεις απασχόλησης με νόημα σε αυτό το παγκοσμιοποίηση ποιημένο πλαίσιο, πώς προσαρμόζονται και εξελίσσονται οι οικονομίες. Οι απαντήσεις σε όλα αυτά είναι πολύ σημαντικές για να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων. Και θέλω να πω και κάτι τελευταίο. Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, τίθεται το εξής ερώτημα, το εξής θέμα. Γνωρίζουμε ότι οι δεξιότητες που διδάσκουμε και τα προγράμματα σπουδών που καταρτίζουμε σήμερα προετοιμάζουν ανθρώπους για θέσεις απασχόλησης που δεν υπάρχουν ακόμα. Και αυτό είναι ο τρόπος, με το, το σημαντικός τρόπος να προβλέψουμε τις ανάγκες. Θα πρέπει δηλαδή να οικοδομήσουμε, να δημιουργήσουμε μια δυνατότητα προσαρμογής. Και αυτό είναι μοναδικό χαρακτηριστικό της χρονικής συγκυρίας της υφιστάμενης και θα πρέπει να επιταχύνουμε, να εντείνουμε τις προσπάθειές μας προς αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστώ η Πρόεδρος. Και εμείς σας ευχαριστούμε. Ο κύριος Μαχτά. Και μετά η κυρία Ρέγνερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Οστίνη, δεν προφέρω σωστά το όνομά σας. Δεν πειράζει. Θέλετε να είστε, φιλοδοξείτε να γίνετε διευθυντής ε, του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και ήρθατε να μας παρουσιαστείτε. Καταρχάς λυπούμε γιατί μιλάτε μπροστά σε τρεις βουλευτές. Είναι πολύ κρίμα αυτό. Και λυπούμε επίσης για αυτά που νιώθω υποχρέωση να σας πω. Μεταξύ ε, των τεσσάρων υπηρεσιών, το SEDEFOP, η ΟΤΣΑ και το Eurofond και το δικό σας το ETF, ε, Τις άλλες τρεις μπορούμε να ανεχθούμε την αξιολόγησή τους. Τις περάσαμε από κόσκινο το τελευταίο 1,5 χρόνο και εγώ θεωρούσα ότι ήδη με τρεις ήταν υπερβολικός ο αριθμός τους, αλλά λυπούμε, θεωρώ ότι το Ίδρυμά σας είναι απαντελώς άχρηστο. Ο μόνος λόγος να είναι κανείς σε αυτή την υπηρεσία είναι για να ασπαταλεί προϋπολογισμό σε χώρες μη ευρωπαϊκές, ε, των οποίων η πολιτική κατάσταση είναι επισφαλής, για να μην μιλήσω για την κατάσταση ασφαλείας. Θέλετε να μιλήσουμε για την Αλβανία, την Ελευκορωσία, την, το Αζερβαϊτζάν, τη Μακεδονία, λέει ο μιλητής, τη Γεωργία, το Ισραήλ, την Ιορδανία, το Κοσφοπέδιο, την Κυργυζία, τη Λιβύη, τη Μολταβία και το Μαυροβούνιο και το Μαρόκο και την Παλαιστίνη και τη Ρωσία και τη Σερβία και τη Συρία, το Τατζικιστάν, την Τινησία, την Τουρκία, το Τουρκμενιστάν, την Ουκρανία ή το Πράγματι είναι αυτά ευρωπαϊκά διακυβεύματα, αυτά που γίνονται εκεί πέρα. Προλίγου κάναμε τον απολογισμό της Συνόδου Κορυφή και του Eurogroup με τον Επίτροπο Ντομπρόφσκι, Στίσεν και Μοσκοβισή, με αυτούς τους επιτρόπους. Και επανειλημμένος έχει υποθεί ότι υπάρχει απόκληση μεταξύ των ε, ε, καταρτήσεων και των προσδοκιών της αγοράς εργασίας. Τα προσόντα δεν αντιστοιχούν σε τίποτα. Το χάσμα και το ρήγμα μόνο βαθαίνει. Και χάρη στο Ίδρυμά σας θα δώσουμε 18 εκατομμύρια ευρώ προϋπολογισμό που θα στραφεί προς άλλες χώρες. Προϋπολογισμό που θα βγει από τις τσέπες των συμπολιτών μας, των Ευρωπαίων πολιτών μας, για τους οποίους εκφράζουμε τη λύπη μας ότι δεν έχουν αρκετή κατάρτιση και εκπαίδευση και θα τα πάρουμε αυτά για να τα δώσουμε στις άλλες χώρες για να αποκτήσουν οι άλλοι. Και πριν θελήσουμε λοιπόν να, συνεχώς να διαδίδουμε διδάγματα και μαθήματα που θα πρέπει να διδαχθούν οι υπόλοιποι, κύριε Διευθυντά, θα ήταν καλό η Ευρωπαϊκή Ένωση με τα χρήματά της να ενδιαφερθεί πρώτα και πάνω απ' όλα για την εκπαίδευση, την κατάρτιση και γενικότερα τα συμφέροντα των Ευρωπαίων πολιτών. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ονεστίνη. Το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα που εδρεύει στο Τωρίνο βεβαίως και έχει ως μέλημά του κύριο να καλλιεργήσει τις σχέσεις και να αναπτύξει σχέσεις εντός του πλαισίου μιας πολύ συγκεκριμένης πολιτικής που είναι η δυνατότητα εξέλιξης και ανάπτυξης ανθρωπίνων χώρων στις γειτονικές χώρες γειτονικέ με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Διακύβευμα δεν είναι να σπαταλήσουμε χρήματα αλλού, αλλά να σταθεροποιήσουμε τη γειτονιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό είναι πρόκληση για όλους μας και κάθε πρόκληση συνεπάγεται κόστος. Εάν δεν έχουμε γείτονε σταθερούς, αν έχουμε γείτονε με αστάθεια, τότε τα προβλήματα έρχονται και στη δική μας ε, αυλή. Σε αυτή τη διαδικασία λοιπόν διεύρυνσης ή συνεργασίας έχουμε συνάψει συμφωνίες συνεργασίας. Δεν είναι όλα στραμμένα προς τη διεύρυνση. Έχουμε υπογράψει συμφωνίες που προβλέπουν συνεργασίες σε πολλαπλά επίπεδα. Το να καταλαβαίνει κανείς καλύτερα τα skills, τις δεξιότητες, τα προσόντα, τον τρόπο με τον οποίο οι χώρες αυτές αξιοποιούν το δυναμικό τους. Το να μπορούμε να το καταλάβουμε αυτό είναι πλεονέκτημα για εμάς στην Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί μπορούμε να εκμεταλλευτούμε, να αξιοποιήσουμε αυτές τις ανάγκες. Οι ανάγκες μας μπορεί να είναι διαφορετικές αλλά μπορεί να είναι και συμπληρωματικές και μας χρειάζεται η εμπειρογνωμοσύνη τους η υπηρεσία δεν προβαίνει σε αλληλοεπικαλύψεις. Έχει δημιουργήσει εμπειρογνωμοσύνη, τεχνογνωσία που είναι πολύ χρήσιμο εργαλείο για τα θεσμικά όργανα και για το ίδιο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στοχοθετούνται καλύτερα οι πολιτικές μας δράσεις. Βρίσκουμε τρόπους συνεργασίες, συνεργασίας με γείτονες που θεωρούμε σημαντικούς. Σημειώνω επίσης ότι πράγματι έχουν υπάρξει αξιολογήσεις της υπηρεσίας και πρόσφατες που οδηγούν στη διαπίστωση τη γενικότερη ότι η υπηρεσία πολύ καλά ε, διαδραματίζει ε, το ρόλο της και επιτελεί τα καθήκοντά της και πρέπει προς αυτή την κατεύθυνση να εντείνουμε τις προσπάθειές μας και συμφωνώ απολύτως. Αυτή η διαπίστωση με βρίσκει σύμφωνο και μάλιστα, σε σχέση με τις λοιπές υπηρεσίες που αναφέρατε, θεωρώ ότι η συνεργασία μαζί τους είναι θεμελιώδης, είναι εξαιρετικά σημαντική. Η σχέση μεταξύ ε, των υπηρεσιών που ασχολούνται με την ανάπτυξη δράσεων ε, εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης και η συνεργασία με την υπηρεσία του Τωρίνου, που αποτελεί και το συνδοτικό με τις πιο σημαντικές γειτονικές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι σημαντικό ε, συγκριτικό μας ε, πλεονέκτημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Ρέγνερ παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Προς τον βουλευτή που έλαβε το λόγο πριν θα ήθελα να πω πως το ETF και το CEDEFOP είναι δύο εντελώς διαφορετικές υπηρεσίες αρκεί να κοιτάξει κανείς τα καθήκοντά τους λίγο πιο κοντά και τότε θα διαπιστώσει τι πρέπει να επιτελέσει το ETF και θα διαπιστώσει πως τα δύο δεν μπορούν να συγκριθούν το ETF βοηθά στην αναχέτηση μεταναστευτικών ροών, επειδή εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση είμαστε πεπισμένοι πω η παιδεία Φυσικά για εμά του πολίτε τη Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά επίση για αυτού που αντιμετωπίζουν μεγάλε δυσκολίε και βρίσκονται εκτό αυτής. Η παιδεία λοιπόν αποτελεί το κλειδί για την αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων. Γι' αυτό και είναι πολύ σημαντικό να κάνει κανεί κάτι προληπτικά και να μην παραπονιέται μόνο όταν δυσκολεύουν τα πράγματα. Η ερώτησή μου προ εσά η έως τώρα διευθύντρια έκανε εξαιρετική δουλειά. Έχετε κάποια ειδικά προσωπικά κέντρα βάρους. Κάτι που σας απασχολεί ιδιαίτερα που θα θέλατε να ενσωματώσετε στην εργασία επιπρόσθετα και έχετε κάποιες χώρες τις οποίες θέλετε να επικεντρώσετε. Ναι, μας δώσατε μια καλή επισκόπηση, γειτονία, ναι, είναι πολύ σημαντικό, αλλά έχετε ίσως επίσης κάποιο πολύ προσωπικό θέμα που θα θέλατε να μεταφέρετε ενδεχομένως στο ETF. Σας ευχαριστώ για το ερώτημά σας. Ως προς την ειδική προσέγγιση και τα επιμέρους θέματα, θεωρώ ότι ως υπηρεσία θα πρέπει να εστιάσουμε το ενδιαφέρον μας στην επίτευξη των στόχων μας. Η ανάπτυξη του ανθρωπίνου κεφαλαίου είναι ε, εμβληματικό σημείο σε ό,τι αφορά την εντολή που έχει δοθεί στην υπηρεσία. Να δώσουμε έμφαση ε, σε αυτά τα οποία μαθαίνουμε εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης για να μπορέσουμε να τα μεταφέρουμε, να τα μεταφράσουμε και να τα ενσωματώσουμε στις σχέσεις με τις τρίτες χώρες. Όλα αυτά πρέπει ε, να ε, λύνονται και να διευθυντούνται στο σημείο από το οποίο πηγάζουν και θέλω να δοθεί έμφαση προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτό που συμβαίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση να μεταλαμπαδεύεται στις τρίτες χώρες και αυτό θα γίνει σε αγαστή συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα λοιπά θεσμικά όργανα και τις λοιπές υπηρεσίες. Νομίζω ότι η Γενική Διευθύντρια της Υπηρεσίας έχει κάνει εξαιρετική δουλειά και μπορούμε να ε, κάνουμε ακόμα περισσότερα μέσω ε, προγραμμάτων ανταλλαγής και θα προσέθετα ότι είναι το σημαντικό, είναι να περάσουμε χρόνο ε, με συζήτηση, με προβληματισμό, με αποκοινού αξιολόγηση για να καθοριστούν τα βασικά στάδια για την ανάληψη δράσης στη συνέχεια. Από εκεί και πέρα, οι κανονισμοί, το, η εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι, ε, συγκροτούν το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα κινηθούμε. Θα πρέπει ενδεχομένως το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης να ε, επικεντρώσει το ενδιαφέρον του σε ορισμένες χώρες που θα αποτελέσουν και ύψιστη προτεραιότητα, τις χώρες τις οποίες μπορεί να φέρει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Οι χώρες που αναφέρατε ε, βρίσκονται σε πολύ διαφορετικό στάδιο ε, η μία από την άλλη σε ό,τι αφορά τις σχέσεις τους με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα έλεγα λοιπόν να στρέψουμε κατά κύριο λόγο το ενδιαφέρον μας στις χώρες με τις οποίες έχουμε στενότερες σχέσεις, γιατί εκεί έχουμε πλειάδα διαθέσιμων εργαλείων, γιατί εκεί υπάρχουν προοπτικές ενίσχυσης της συνεργασίας. Ε, μιλούμε για τις χώρες που είναι υποψήφιες για μελλοντική διεύρυνση, ή μιλούμε για τις χώρες με τις οποίες έχουμε ειδικέ συμφωνίες συνεργασίες για τις χώρες που τις βοηθούμε στις μεταβατικές περιόδους που διανύουν. Αυτά πρέπει να είναι προτεραιότητά μας. Όλα αυτά αλλάζουν πολύ γρήγορα. Αυτό συμβαίνει στις σχέσεις και πρέπει να κρατήσουμε δυνατότητες ε, μεταφοράς τεχνογνωσίας για τις χώρες που βρίσκονται στον κατάλογο χωρών χαμηλότερης προτεραιότητες. Γιατί μπορεί κάτι να αλλάξει, θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι και να διατηρήσουμε το επίπεδο τεχνογνωσίας μας. Νομίζω ότι μόλις καταλήξουμε στις βασικές προτεραιότητες για τις ε, κοντινές μας χώρες, θα πρέπει να δουλέψουμε για να διατηρήσουμε το ίδιο επίπεδο τεχνογνωσίας και για τις υπόλοιπες που ε, είναι στη σειρά. Η Πρόεδρο, σας ευχαριστώ. Ο κύριος Μπέκερ θέλει να θέσει ερωτήματα. Παρακαλώ. Uh, Γεια σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καθώς δεν ήμουν παρόν κατά την ομιλία, δεν θα ήθελα να επισέλθω σε λεπτεμέρειες, επειδή έχουμε μια γενική άποψη, στο πλαίσιο της οποίας θα ήθελα να ρωτήσω την, ερ... ερώτησή μου. Ποιες θα είναι οι μεγαλύτερες προκλήσεις στην πολιτική αυτή και ποια θα πρέπει να είναι τα επόμενα βήματα για να επιτευχθούν δεξιότητες στις αναπτυσσόμενες χώρες. Τώρα ξέρω, έχει ήδη απαντηθεί, οπότε δεν θέλω να ενοχλήσω τους υπόλοιπους. Εάν η αγαπητή συνάδελφος θέλει, είναι το κατάλληλο αποτέλεσμα της συνεδρίασης αυτής. Ευχαριστώ. Ευχαρίστως μπορώ να δώσω μια σύντομη σύνοψη. Η μεγάλη πρόκληση είναι η παγκοσμιοποίηση και πώς θα προσαρμοστούμε σε αυτήν, πώς θα χρησιμοποιήσουμε τα εργαλεία και τις δεξιότητες που αναπτύσσουμε ως Ευρώπη για να προσαρμόσουμε επίσης τους γείτονές μας ώστε να έχουμε μια σταθερή γειτονία. Αυτή είναι μια πολύ σύντομη σύνοψη. Ευχαρίστω αργότερα μπορούμε να συζητήσουμε αν χρειάζεστε κάποιες περισσότερες πληροφορίες. Συνάδελφε Γκέρικε, έχετε κάποια ερώτηση. Ωραία. Ήταν πολύ σύντομη και αποδοτική η σημερινή συνεδρίαση, θα έλεγα. Υπάρχει κάτι που θέλουμε να προσθέσουμε πριν αφήσουμε τον κύριο Ονεστίνη να πάει να πάρει το μισθωτιανό του ίσως. Υπάρχει κάτι που θα έπρεπε να, έχουμε ρωτήσει, να σας έχουμε ρωτήσει και δεν ρωτήσαμε. Ρωτήσατε τις τέλειες ερωτήσεις, απάντησε ο κύριος Ανεστίνη. Οπότε δυσκολευόμαστε ακόμα περισσότερο να βρούμε κάποια επιπλέον ερώτηση ή να θέσουμε κάποια απρόβλεπτη ερώτηση, αλλά είμαστε λίγοι εδώ. Και πιστεύω πως πρέπει να διακόψουμε εδώ. Είχαμε μια καλή συζήτηση, δεν ήμασταν πολύ σκληροί. Ακούσαμε τα πιο σημαντικά ζητήματα για μας, λάβαμε απαντήσεις σε αυτά, ακούσαμε, αποκτήσαμε μια εικόνα των αξιών και των επιθυμιών σας, όπως και των φιλοδοξιών σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε. Και τώρα μπορούμε να παραμείνουμε εδώ για μια σύντομη συζήτηση μετά την αποχώρησή σας. Ο Νεστίνη, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω. Προσδοκώ με χαρά τη συνεργασία με την Επιτροπή αυτή και το Κοινοβούλιο και είμαι σίγουρος ότι πρόκειται για την αρχή μιας πολύ καλής συνεργασίας. Ευχαριστώ.